Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Καλωσορίζω τους παρόντες και τους εξαποστάσεως ε, συνδεόμενους. Ελπίζω να περάσετε καλά στις διακοπές και ελπίζω και εσείς και οι οικοί σας να χαίρουν άκρας υγείας. Γιατί ακόμη χαλεποί καιροί συνεχίζονται. Πάμε κατευθείαν στην ημερήσια διάταξη. Πρώτα να την εγκρίνουμε. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, εγκρίνεται σε διάταξη. Δεν βλέπω αντιρρήσει. Σε ό,τι αφορά τι ανακοινώσει του Προέδρου, ε, σημείο 2. Η πρώτη, ο πρώτος γύρος ψηφοφορίας θα γίνει μεταξύ 15 και 45 και 16 και 45 και αύριο μεταξύ 14 και 45 και 16 και 45. Όσοι ε, λάβουν μέρος ε, στην ψηφοφορία, είτε από την αίθουσα είτε εξ πρέπει να χρησιμοποιήσουν το σύστημα της αποστάσεως ψηφοφορίας. Έχουμε διερμηνία στα γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πολωνικά, πορτογαλικά και κροατικά. Και επειδή έχουμε διερμηνία είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε αυστηρά το χρόνο γιατί αλλιώς θα χάσουμε τη διερμηνία αν υπερβούμε το χρόνο μας. Σημείο 3. Η ετήσια μας συνεδρίαση με τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μάλιστα αυτή τη φορά θα είναι διαφορετική η συνάντηση που θα έχουμε με προσώπους αποκεντρωμένων οργανισμών, γιατί ε, θα ε, εξετάζουμε συνήθως ε, τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τις περικοπές που πρότεινε το Συμβούλιο. Αυτή τη φορά όμως είμαστε σε λίμπο ακόμη, κάπως μετέωροι, γιατί δεν έχουμε ακόμη ένα σταθερό χρηματοδοτικό πρόγραμμα ή τα τελικά ποσά για τις δημοσιονομικές προοπτικές. Θα ζητήσουμε όμως τον αντίκτυπο Τη κρίση του κορονοϊού και πώ επηρεάζει του οργανισμού. Καλωσορίζουμε τον κύριο Χάνζεν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων που εδρεύει στο Ελσίνκι και εκπροσωπεί μάλιστα το δίκτυο των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Χάνσεν, θα μας ενημερώσετε για τον προβληματισμό και τι προοπτικές των οργανισμών. Μόνο εύκολο δεν είναι το έργο σας ε, δεδομένων των συνθηκών δεν μπορείτε να κάνετε προγραμματισμό για, ούτε καν για μονοετή κύκλο εργασία, για να μην πω για πολυετή. Και μια και εκρεμούν οι διοργανικές διαπραγματεύσεις από δημοσιονομικής πλευράς, είστε και εσείς περιορισμένοι ως προς τον προγραμματισμό σας. Κύριε Χάνσεν, έχετε ένα τέταρτο περίπου για να μας κάνετε την παρουσίασή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμη... Ευρωβουλευτέ της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θα ήθελα το δεκάλεπτο τέταρτο που έχω στη διάθεσή μου να σας περιγράψω καταρχήν το έργο του δικτύου των οργανισμών, να σας μιλήσω για τα επιτεύγματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη διάρκεια της κρίσης COVID-19 και να σας μιλήσω λίγο και για τις στρατηγικές μας προοπτικές και τι ανάγκη έχουμε ως δίκτυο να αναλάβουμε μια στρατηγική δράση. Το δίκτυό μας, το δίκτυο οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εθελοντικό και καλύπτει 48 οργανισμούς και ε, κοινέ συμπράξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με, επαναλαμβάνω, εκούσια εθελοντική συμμετοχή. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι μέσω ενισχυμένης συνεργασίας να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον αντίκτυπό μας και ε, να κάνουμε ανταλλαγή γνώσεων προκειμένου να εξυπηρετήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά. Και για να σας περιγράψω πώς λειτουργεί το δίκτυό μας και εξετάζοντας τις προκλήσεις αλλά και τα επιτεύγματα μας στη διάρκεια της κρίσης ε, του COVID-19, είναι χαρακτηριστικό το πώς δράσαμε για το πώς αντιλαμβανόμαστε το έργο μας. Μέριμνά μας είναι να προστατεύσουμε το μέλλον μας. Να έχουμε μέλλον δηλαδή, πρώτα απ' όλα. Και μία από τις, από αδερφούς οργανισμούς, η, οργανισμός, το Κέντρο Ελέγχου Πρόληψης των Νόσων, βρέθηκε στο επίκεντρο του έργου και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη προσπάθησε να αντιμετωπίσει την κρίση. Αλλά και το δίκτυο έδωσε μια πλατφόρμα και εξασφάλισε την καλή συνεργασία του Κέντρου Πρόληψη των Νόσων με τους άλλους οργανισμούς, ώστε να έχουμε άμεση δράση για ευρωπαϊκά οριζόντια ζητήματα που έχριζαν μια πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση. Και δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτή τη συνεργασία και τη συζήτηση που είχαμε ήταν οι συζητήσεις με τον οργανισμό των μεταφορών με, τον, με το κέντρο πρόληψης νόσου. Προσπαθήσαμε να δούμε πώς ο οργανισμός για τις μεταφορές μπορεί να αντιμετωπίσει ε, την κρίση. Επίσης, ε, συνεργασία με την Ρωσία από τον Οργανισμό για την Επαγγελματική Υγεία και εκεί φροντίσαμε να αντιμετωπίσουμε την πανδημία στο χώρο εργασίας. Επίσης, με την υποδομή του δικτύου μας, επιτρέψαμε στους ε, διάφορους αυτούς οργανισμούς που σας ανέφερα να έχουν πιο άμεση και ταχεία συνεργασία. Ένα άλλο παράδειγμα είναι ότι το δίκτυό μας πολύ γρήγορα σύστησε μια ομάδα κρούσης των οργανισμών για να αναπτύξει σαφείς συγκεκριμένες προτάσεις που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι οργανισμοί για να αντιμετωπίσουν ο καθένας στον τομέα του την κρίση COVID. Για παράδειγμα, είχαμε συνεντεύξεις ε, online μέσω του διαδικτύου και εξετάσαμε τις διάφορες ε, φάσεις ε, και τα διάφορα στάδια για να επιστρέψουν να επιτρέψουμε την τηλεεργασία και μετά την επαναφορά στο χώρο εργασίας. Γενικώ συζητήσαμε πολλές τέτοιες προκλήσεις της κρίσης και αυτά ήταν δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς το δίκτυο ενισχύει την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί επαναλαμβάνω διευκολύνει την ε, αμεσότερη και στενότερη συνεργασία. Βέβαια, όπως όλοι, αντιμετωπίσαμε και προκλήσεις ε, όλα τα θεσμικά όργανα και όλοι οι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξαν προβλήματα με την εκτέλεση του προπολογισμού του 2020 έγιναν και κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα εργασίας ε, σε αρκετούς οργανισμούς. Πάντως, γενικώ καταφέραμε να ανταποκριθούμε και να ανταπεξέλθουμε στην αποστολή μας. Βέβαια, οι μακροπρόθεσμη συνέπεια της κρίσης COVID δεν είναι ακόμη σαφείς. Πάντως, συνεργαζόμαστε με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, αλλά περιμένουμε την οριστικοποίηση του προπολογισμού. Υπάρχουν κάποια προβλήματα στις προσλήψεις και στις προμήθειες. Εμείς έχουμε προσλάβει προσωπικό ακόμη και στη διάρκεια της κρίσης. Και ξεκινήσαμε την απασχόλησή τους με τηλεεργασία φυσικά, γιατί δεν μπορούσαν να μεταβούν στον χώρο εργασίας τους και στον τόπο εργασίας τους. Υπήρξαν και κάποια προβλήματα, κάποιοι στενόποι. Και επίση, ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να κάνουμε πιο ελαστική χρήση και των ανθρώπινων και των χρηματοοικονομικών μα πόρων. Τέλο, ε, μακροπρόθεσμη οργάνωση, ε, θέματα κοινωνική συνοχή και συνεργασία. είναι θέματα κουλτούρα ουσιαστικά των οργανισμών, των οργανισμών μας, αλλά αυτό είναι ένα κοινό θέμα που συμμερίζονται και άλλα θεσμικά όργανα, για να μην πω ο μισός κόσμος. Αυτά ήταν κάποια παραδείγματα των επιτεγμάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε και το πώς μπορεί το δίκτυο να μας βοηθήσει και να εδραιώσουμε τα επιτεύγματα και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Τώρα κάποιες πιο στρατηγικές προοπτικές. Φυσικά δημιουργήθηκε μια νέα κανονικότητα με την κρίση COVID που θα την αντιμετωπίσουμε και σε συνεργασία μαζί σας και μόνοι μας ξεχωριστά ο κάθε οργανισμός η επταετή στρατηγική ανταποκρίνεται και στα δημοσιο... στις δημοσιονομικές προοπτικές και αυτό ισχύει για όλο το δίκτυο των οργανισμών και επιμέρους τομείς, καινοτομία, βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση και προσπαθούμε εμείς μέσω του δικτύου και χάρη ε, στις δεξιότητες των οργανισμών προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε μια πιο μακροπρόθεσμη στρατηγική. Επίσης, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γίνουμε υπόδειγμα διοικητικής αριστείας. Όχι μόνο οι μεμονωμένες, οι μεμονωμένοι οργανισμοί, αλλά και στη διαρθρωτική μας συνεργασία μέσω του δικτύου. Θέλουμε να γίνουμε υπόδειγμα, παράδειγμα προς μίμηση διοικητικής αριστείας. Επίσης, έχουμε συνεργασία αξιοποιώντας πολλά εργαλεία. Προσπαθούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και με τα εργαλεία αυτά να υλοποιήσουμε το, σχέδιο, το πρόγραμμα εργασιών μας και να αξιοποιήσουμε τα θετικά στοιχεία προσπαθώντας να αντισταθμίσουμε τα αρνητικά στοιχεία, τα πιο αδύναμα σημεία. Αυτή είναι μια φιλοδοξία βασική της επταετούς μας στρατηγικής. Επίσης θέλουμε να τηρήσουμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ένα νέο ψηφιακό πράσινο κόσμο και τη μετάβαση σε μια οικολογική, φιλοπεριβαλλοντική και πιο βιώσιμη οικονομία. Και για παράδειγμα ο δικός μου οργανισμός των χημικών προϊόντων ε, το Διοικητικό μας Συμβούλιο ανέλαβε την ε, δέσμευση μέχρι το 2030 να γίνουμε κλιματικά ουδέτερος οργανισμός. Γιατί και μέσω της Νέας Πράσινης Συμφωνίας οι οργανισμοί αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Έτσι και ως οργανισμός μεμονωμένος και ως δίκτυο συμβάλλουμε να, στην υλοποίηση των κοινών ευρωπαϊκών στόχων με τη συνεργασία και το έργο μας. Επίσης, θέλουμε να παραμείνουμε ένας αξιόπιστος και πολύτιμος θεσμικός εταίρος και ως δίκτυο και μέσω του δικτύου να υλοποιήσουμε το βασικό μας στόχο, να στηρίξουμε δηλαδή την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη και τα κοινοτικά θεσμικά όργανα, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και για να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τηρήσουμε δύο προϋποθέσεις, όλοι οι οργανισμοί. Καταρχήν, αυτό που λέμε ελαστικότητα, ευελιξία. Και μια άλλη προϋπόθεση ε, θα αφορά την ανάληψη νέων καθηκόντων και αποστολών. Σε ό,τι αφορά την ελαστικότητα, όταν λέμε ότι θέλουμε ελαστικότητα, εννοούμε ότι θέλουμε περισσότερη ελαστικότητα, περισσότερη ευελιξία και στον τρόπο χρηματοδότησης, αλλά και στον τρόπο στελέχωσης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού μας. Και δεν θέλουμε ελαστικότητα μόνο για να είμαστε πιο ικανοποιημένοι. Θέλουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα για να μπορέσουν οι οργανισμοί που είναι κοντά στην Ευρώπη και κοντά στους πολίτες, για να μπορέσουν να εφαρμόσουν καλύτερα την πολιτική τους, να μπορούν να κατανείμουν τους πόρους τους ταχύτερα. Γιατί εμείς λαμβάνουμε πόρους, κατανέμουμε πόρους και όταν ε, ολοκληρώνεται μια αποστολή στερούμαστε για κάποιους πόρους. Οπότε χρειάζεται ελαστικότητα και στη χρηματοοικονομική πλευρά, αλλά και στην ε, πλευρά της στελέχωσης των οργανισμών. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις μελλοντικέ μας προκλήσεις. Ένα από τα παραδείγματα μας δείχνει η κρίση COVID. Για παράδειγμα, το κέντρο πρόληψης νόσου, αλλά και ο οργανισμός φαρμάκων, είχαν αύξηση του φόρτου εργασίας και ο οργανισμός φαρμάκων. Θέσπισε ένα ολόκληρο πρόγραμμα για την ε, ανακάλυψη εμβολίων κατά του κορονοϊού. Ε, υπήρξε μια μεγάλη αύξηση του φόρτου εργασίας των δύο οργανισμών ε, κάτι που δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν με αντίστοιχη στελέχωση. Ούτε με τη μετάθεση από τον ένα οργανισμό στον άλλο καλύπτονται κάποια κενά. Θέλουμε μεγαλύτερη ελαστικότητα στον τρόπο της στελέχωσης. Επίσης, ξέρουμε ότι ο οργανισμός για τον έλεγχο πρόληψης και των νόσων, πρόληψη και ελέγχου των νόσων, είχε τεράστια αύξηση του φόρτου εργασία. Γι' αυτό και χρειάστηκε κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση. Είδαμε και με τη μεταναστευτική κρίση. υπήρξε μια διοικητική ακαμψία που εμπόδισε τους οργανισμούς να υπηρετήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο παράδειγμα αυτής της ανάγκης ελαστικότητας προέρχεται από τον Οργανισμό για την Πολιτική Αεροπορία. Αλλά είναι κάτι αντίστοιχο το βιώνουμε και εμείς, στην Οργανισμό Χημικών Φραγμάτων, Χημικών Προϊόντων. Φυσικά υπήρξε μεγάλη απώλεια εισοδήματο στον Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας λόγω της μείωσης των πτήσεων. Θα πρέπει λοιπόν το σύστημα της στάθμισης που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει πιο ελαστικό, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ανελαστικό, άκαμπτο και δεν μπορεί να εξασφαλιστεί συνέχεια δεδομένων των ενωσιαθικών Αυτά ως προς την ελαστικότητα. Τώρα, για τα νέα μας καθήκοντα, αν αναλάβουμε νέα καθήκοντα θα πρέπει να εξοπλιστούμε με τους απαραίτητους πόρους για να ανταπεξέλθουμε. Ή αν δεν έχουμε αρκετούς πόρους για να αναλάβουμε τα νέα μας καθήκοντα, αναπόφευκτα θα πρέπει κάποιες τωρινές μας δραστηριότητες να τις υποβαθμίσουμε στην ιεραρχία των προτεραιοτήτων μας. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε και θα ανταπεξέλθουμε στο φόρτο εργασία. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμό, ένα τέριασμα των πόρων με τα νέα καθήκοντα. Κάτι που διοικητικά δεν είναι πάντα εύκολο. Αυτά λίγο πολύ ως προς την ελαστικότητα και τα νέα μας καθήκοντα. Αυτά είναι προϋποθέσεις για να καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε στο έργο μας και οι μεμονωμένοι οργανισμοί και το δίκτυο. Γνωρίζουμε ότι απαιτεί πολλά από εμά η Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να συμβάλλουμε στην προστιθέμενη ευρωπαϊκή αξία. Και γι' αυτό και οι οργανισμοί και το δίκτυο χαιρόμαστε πολύ που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και προσβλέπουμε στη συνέχιση της αγαστής μας συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάνσεν. Ο κύριος Herbst, Ελκ, που είναι μόνιμος εισηγητής μας για τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Herbst. Με φοβερή αντίχηση όμως. Mr. Herbst, could you please use a headset while... Κύριε Herbst, μπορείτε να δοκιμάσετε πάλι γιατί ο ήχος που φτάνει στην αίθουσα είναι πολύ κακός. Mr. Herbst, please press the speak button. Πιέστε το κουμπί ομιλία παρακαλώ, κύριε Χέρψ. Ναι. Με ακούτε? Λοιπόν, προσπαθώ και πάλι. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο. Δεν φτάνει ο χρόνος για να ευχαριστήσουμε όλους τους οργανισμούς για το εξαιρετικό τους έργο και κάτω από δύσκολες συνθήκες μάλιστα. είναι δύσκολη καιρή πράγματι. Και άλλοι οργανισμοί έχουν πολύ καλές επιδόσεις και γι' αυτό και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους. Τώρα η νέα γενιά αυτό που κάνει είναι ότι μας δίνει την ευκαιρία να στηρίξουμε καλύτερα, the new generation δηλαδή, και να υποφεληθούμε από πολλές ευκαιρίες που προσφέρονται. Και αυτό είναι ευτυχές. Τώρα, συγκρίνοντας τις ανάγκες των οργανισμών για την επόμενη επταετία, η σημερινή πρόταση δεν διασφαλίζει την ικανότητά τους να φέρουν σε πέρας το έργο τους την επόμενη επταετία. Χρειάζονται συνεπώ προτεραιότητες και θα αναγκαστούν να θέσουν και κάποιες αρνητικέ προτεραιότητες και κάποια από τα καθήκοντά τους και οι αρμοδιότητές τους δεν θα έρθουν σε πέρας μέσα στην επόμενη επταετία έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Να κάνω κάποιες παρατηρήσει τώρα, ακόμα, επειδή έχουμε λίγο χρόνο. Νομίζω ότι πολλέ δραστηριότητε οργανισμών για το ίδιο τρίμηνο του 2020 αναβλήθηκαν για το τέταρτο τρίμηνο. Θα δούμε βέβαια πώς θα πάει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν σίγουρα πολλοί περιορισμοί και ίσως αναγκαστούν να προχωρήσουν και σε παραπάνω ακυρώσεις ε, καθηκόντων τους και δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τον προπολογισμό όπως πρέπει. Ελπίζω να μας βοηθήσουν οι οργανισμοί με τις προτεραιότητές μας. Φαίνεται ότι το προσπαθούν, καινοτομία, αηφορία, για μας η διαφάνεια αποτελεί στοιχείο κλειδί για να ξέρουμε πώς δαπανώνται τα κονδύλια ακριβώς. Είμαστε Επιτροπή Προπολογισμών και από τη φύση μας πρέπει να ε, το κοιτάμε αυτό το πράγμα και να ξέρουμε τι γίνεται και να συνδέουμε πάντα τη χρήση των πόρων με συγκεκριμένες δραστηριότητες. Ε, το θέμα των προτεραιοτήτων και η πανδημία δεν πρέπει να είναι σε βάρος άλλων ε, δραστηριοτήτων και σίγουρα προστίθονται και νέε προκλήσει όπω είναι το COVID-19 και όπω είναι βέβαια και η Πράσινη Συμφωνία. Ευχαριστώ και πάλι όλου του οργανισμού για το εκπληκτικό του έργο κάτω από δύσκολε συνθήκε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Γκουεμίνη από τους σοσιαλδημοκράτες, αλλά σας παρακαλώ όλους 1,5 λεπτό να μιλάτε, όχι παραπάνω, για τελειώ δεν θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα με την οργάνωση. Η κυρία Γκουαλμίνη τώρα έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Με ακούτε? Καλώ, Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Χάνσεν για την πλήρη παρουσίασή του και πρέπει να πω επίσης ότι ως δίκτυο και εσείς κάνετε εκπληκτική δουλειά και κάτω από δύσκολες συνθήκες εννοείται. Σας ευχαριστώ πολύ. Και λαμβάνουμε η υπόψη μας το έτοιμά σας για περισσότερη ευελιξία στη χρήση και στην κατανομή των πόρων, προκειμένου να μπορέσετε να ανταποκριθείτε πιο γρήγορα και πιο εύκολα στις ανάγκες και στις απαιτήσεις των πολιτών ο κάθε οργανισμός στον τομέα του έχω κάποιες σύντομες ερωτήσεις. Πρώτον, δεδομένου ότι το COVID βρίσκεται στην κοινωνία μας και θα βρίσκεται και τα επόμενα χρόνια από ό,τι φαίνεται, πιστεύετε ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη Ασθενειών και τον Έλεγχο Ασθενειών διαθέτει αρκετούς πόρους για τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού Πώς πιστεύετε ότι θα τα καταφέρει για να αντιμετωπιστούν ασθένειες όπως αυτή. Επίσης, τα τελευταία χρόνια και για τον επόμενο χρόνο το σχέδιο προπολογισμού προβλέπει μία αύξηση, διακόπτεται η ομιλήτρια, κόβεται η σύνδεση. Δεν υπάρχει σύνδεση με την ομιλήτρια. And finally... Τέλος, υπάρχει πάλι σύνδεση. Η υπηρεσία περιβάλλοντος, ο οργανισμός περιβάλλοντος, πώς θα μπορούσε να συνεισφέρει για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Πώς πιστεύετε ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Στεφανούτα τώρα από το Ρινιού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Στεφανούτα. Ο, κύριο Στεφανούτα. we can hear you but we see. Μπορούμε να σας ακούσουμε, αλλά δεν σας βλέπουμε. Go ahead. Go ahead. Okay. Well,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 Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα αγαπητοί συναδελφοί. Ευχαριστούμε κύριε Χάνσεν. Σας ευχαριστώ για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Φέτος η θέση των οργανισμών είναι δύσκολη. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα για τον προπολογισμό του 2021 ε, και λόγω των απόψεων του Συμβουλίου ορισμένοι προπολογισμοί των αποκεντρωμένων οργανισμών έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, ας δούμε, ε, που αυξήθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως η Frontex, όπου περάσαμε από 137 εκατομμύρια το 2015 σε 322 εκατομμύρια το 2020, με αποτελέσματα αμφισβητήσιμα, θα έλεγε κανείς. Τα ποσά αυτά θα πρέπει να συγκριθούν με τον διορθωτικό προπολογισμό ε, που είχαμε το τελευταίο χρόνο για την Τουρκία με 400 εκατομμύρια και παραπάνω. Αντιλαμβάνομαι την αντιμετώπιση της σημερινής κρίσης που απαιτείται αύξηση ε, κονδύλιων για βοήθεια προς τις ε, χώρες και για διάφορες πληρωμές. Ωστόσο, η ύπαρξη των οργανισμών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει πολλά ερωτήματα. Η βοήθεια του σε επιστημονικό και τεχνικό επίπεδο είναι αμφίβολο τα τελευταία χρόνια, διότι σήμερα έχουμε 6.000 ανθρώπους με υψηλότερο προπολογισμό για την περίοδο 2014-2020. Έχω λοιπόν δύο ερωτήσεις. Μπορείτε να μας πείτε αν στην παρούσα φάση προβλέπονται και η δημιουργία και άλλων αποκεντρωμένων οργανισμών με διεύρυνση αρμοδιοτήτων ε, της κοινότητας ε, σε διάφορους τομείς. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και η δεύτερη ερώτηση η διακυβέρνηση αυτών των οργανισμών πώς θα γίνει και όσον αφορά το κόστος τους, διότι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου λένε ότι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί πρέπει να υφίστανται σε ανώτατες σε κατώτερο επίπεδο από ό,τι προτείνει η Κομισιόν, που σημαίνει μείωση προπολογισμού για τα ε, περισσότερε ενότητες. Οπότε υπάρχουν αφιβολίε για τον προπολογισμό 2021, διότι αναμένουμε την θέση του Συμβουλίου ακόμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Λαπόρτο. Δεν έχουμε λάβει ονόματα από το ECR και την ΚΟΕ. Α, ναι, συγγνώμη. Κυρία Χάρμ, παρακαλώ. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Μπορείτε να με ακούσετε και να με δείτε, ελπίζω, κύριε Χάν. Κύριε Χάν, Χάνσεν, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σας. Αγαπητοί συναδελφοί, οι οργανισμοί κάνουν μια πολύ σημαντική δουλειά. Είναι λοιπόν σαφές ότι θα πρέπει να πρικοδοτηθούν με επαρκή σε οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν όλα τα σημαντικά καθήκοντα που έχουν, τα οποία αυξάνονται και σε αριθμό. Γι' αυτό εμείς οι πράσινοι πιστεύουμε ότι οι οργανισμοί θα πρέπει να λάβουν μεγαλύτερη χρηματοδότηση τουλάχιστον να καλύπτονται τα αιτήματά τους. Και θέλω ειδικότερα να εκφράσω την υποστήριξή μας για καλύτερη και καλύτερη και περισσότερη ε, χρηματοδότηση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Περιβάλλοντος και για τους οργανισμούς που άπτονται της δικαιοσύνης και των ιστορικών υποθέσεων και για την Πράσινη Συμφωνία και τον Κλιματικό Νόμο της Ευρώπης η, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος θα έχει περισσότερα καθήκοντα στο μέλλον. Μπορεί να ε, τελείσει και ως γραμματέας ε, ε, για το μελλοντικό Συμβούλιο Περιβάλλοντο. Γι' αυτό η ΕΕ πρέπει να έχει περισσότερου πόρου, επαρκεί πόρου. Χρειαζόμαστε περισσότερο μόνιμο προσωπικό για καλύτερη περιβαλλοντική παρακολούθηση, ανάλυση δεδομένων και παρακολούθηση. Και για του οργανισμού δικαιοσύνη και εσωτερικών υποθέσεων πρέπει να αυξήσουμε τη χρηματοδότηση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που σε εποχέ σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ακόμη και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, επιτελεί πολύ σημαντικό έργο και το εκτιμάμε. Τέλο, η αύξηση τη χρηματοδότηση για τη Eurojust θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Στο μέλλον, ο οργανισμό αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο για την πρόθεση τη πρόσβαση στη δικαιοσύνη, κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Προσδοκώ να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε σε αυτά τα σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Χάν. Όπως είπα, δεν μας έχει δώσει ομιλητές ούτε το ΕΣΥΑΡ, ούτε η ΓΚΟΕ, ούτε η μη εγγεγραμμένη. Έχει αλλάξει αυτό. Διαφορετικά, κύριε Τζόντσα. Ο κύριος Τζόντσα. Θα είμαι, θα είμαι λακωνικό. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα. Σίγουρα οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί είναι αποκεντρωμένοι και σίγουρα οι οργανισμοί θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση την αποτελεσματικότητά τους και το κατά πόσο ανταπεξέρχονται στα καθήκοντά τους. Και πολλοί μας ρωτάνε πόσα κονδύλια και γιατί ε, ανατίθενται στους οργανισμούς. Γιατί είναι διαφορετική λειτουργία των οργανισμών. Οι περισσότεροι βέβαια οργανισμοί λειτουργούν ε, σωστά και αποτελεσματικά. Αλλά όταν ε, εντοπίζουμε λάθη θα πρέπει να τα διορθώνουμε για να αποδείξουμε ότι έχει νόημα η σύσταση, ίδρυση στον οργανισμό και είναι πραγματικά επιτυχημένη. Σίγουρα ε, είναι σωστή αποτελεσματική και θα πρέπει να είναι και χρηστή η διαχείριση και να στελεχώνονται με πραγματικούς επαγγελματίες. Αξιολογούμε λοιπόν θετικά την ε, λειτουργία πολλών οργανισμών, αλλά θέλουμε πιο αυστηρό έλεγχο όλων των οργανισμών, γιατί μερικές φορές ε, δεν ε, είναι απόλυτα χρηστή η διοίκησή και θα πρέπει να το εξετάζουμε. Ευχαριστώ κύριε Τζοντσό. Δεν υπάρχει ομιλητής από την ΚΟΕ. Πάμε στον κύριο Κουλακούσιτς, ε, Μία εγγεγραμμένος. Σα ευχαριστώ. Όπω είπε και ο προλαλής σας, το κλειδί για τη χρηματοδότηση των αποκεντρωμένων οργανισμών θα πρέπει να είναι η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητά τους. Ε, διαβίουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση που προκλήθηκε από μια πανδημία, από μια μεταδοτική νόσο, από μια λίμωξη. Κατά τη γνώμη μου, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου των Νόσων μας απογοήτευσε ποιος, ποιο είναι το αποτέλεσμα των εργασιών αυτού του οργανισμού. Τι χρήσιμο ακούσαμε από αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου για να αξιολογήσουμε την επικινδυνότητα της πανδημίας. Τίποτα δεν ακούσαμε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου, σαν να μην ε, υπήρξε η πανδημία. Είναι πραγματικά ε, κομικοτραγικό ε, να βρίσκεται έδρα της ε, του κέντρου πρώιμης στη Σουηδία να σταματήσει ε, να λειτουργεί και ε, να μην δίνει κανένα λόγο για, το, για την πανδημία. Κατά τη γνώμη μου, το Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου δεν αξίζει κανένα απολύτω κονδύλιο και χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Χάνσεν, για αυτή την παρουσίαση. Όπως γνωρίζουμε όλοι, συχνά οι οργανισμοί έχουν λειτουργικό ρόλο. Ε, μπαίνουν στην πραγματική δράση. Θα ήθελα να αναφερθώ ειδικότερα σε διάφορους οργανισμούς ε, στον τομέα των ε, πολιτικών ελευθεριών, του ασύλου, της μετανάστευσης και του κράτους δικαίου. Ανισχώ και εγώ, όπως διάφοροι συνάδελφοι, όσον αφορά τις συνέπειες των αποφάσεων του Συμβουλίου που προτείνουν ε, ακόμα μεγαλύτερη μείωση του προπολογισμού των οργανισμών, αν σκεφτεί κανεί ε, τι προοπτικέ που έχουμε μπροστά μα. Α σκεφτούμε για παράδειγμα την Ευρωπόλ. Η αποστολή τη ε, κατά την κρίση του COVID υπήρξε ουσιαστική, διότι βοήθησαν να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα σε αστικό επίπεδο, ε, συγγνώμη, σε online. Να σας υπενθυμίσω έναν αριθμό. Η παιδική πορνογραφία διπλασιάστηκε στους τρεις μήνες του αποκλεισμού αυτού όσον αφορά την κυκλοφορία ε, παιδικής πορνογραφίας online. Πρέπει λοιπόν να αυξηθούν οι δυνατότητες, τα μέσα που δίνουμε σε αυτόν τον οργανισμό, ούτως ώστε να μπορεί να επιτηρεί σωστά και να εφαρμόζει σωστά τον κανονισμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ευρωπόλ ε, χρειάζεται παραπάνω προπολογισμό και προσωπικό. Ε, ας δούμε μετά τον ε, Ευρωπαϊκό Εισαγγελέα, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, την Eurojust που ανέφεραν οι συναδελφοί μου. Ανησυχούμε λοιπόν όσον αφορά το κατά πόσο θα έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν στόχους που ωστόσο έχουν οριστεί για αυτούς τους οργανισμούς. Τέλος, όσον αφορά το άσυλο και τη μετανάστευση, τομεί με πολλές δυσκολίες και πολλά προβλήματα και πολλούς προσανατολισμούς ε, που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο στο πλαίσιο της εντολής της κυρίας Φαντερ Λάιεν, όσο και στο πλαίσιο ανακοινώσεων που έγιναν στο σχέδιο ανάκαμψης. Είναι πολύ σημαντική η αύξηση των μέσων για την Frontex, για το ίδιο e Λίσα, για την ΕΑΣΟ ώστε να μπορέσουν να διασφαλίσουν ε, ότι θα επιτευχθούν οι φιλοδοξίες ε, για έλεγχο της μετανάστευσης με μέσα εφαρμοσμένα και ελεγμένα. Αυτή είναι πρωταρχική αποστολή των οργανισμών αυτών. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε τα απαραίτητα μέσα για να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Χώσικ από το Ρινιού. Uh, I would like to in more detail about... Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο πιο λεπτομερώς για έναν οργανισμό, αν μου το επιτρέπετε. Για τον ΕΚΑ που ε, από τη φύση του έχει κάποιους πιο ψηφιακούς, κάποιους πιο πράσινους στόχους και αναρωτιέμαι τι γίνεται για τους τομείς πολιτικής. με το περιεχόμενο το ότι πρέπει να επιτευχθεί και τέλος όσον αφορά τους πόρους. Η ευελιξία για τα ποσά, η σταθερότητα των ποσών αυτών, πώς θεωρείτε ότι θα είναι όσον αφορά τους διαθέσιμους πόρους, ούτω ώστε να υποστηριχθεί σωστά η υλοποίηση των πολιτικών. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Χάνσεν, αυτές ήταν οι παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών είτε στην αίθουσα είτε εξ αποστάσεως, οπότε σας ακούμε τώρα για τις απαντήσεις σας. Ο κύριος Χάνσεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους τους αξιότιμους ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω κάπως συνοπτικά και μετά θα σας πω σε ποιες δεν έχω απαντήσει και πώς θα πάρετε τις απαντήσεις σας μετά. Λοιπόν, ξεκινάω με το εξή. Πρώτα απ' όλα, θέλω να σας καθησυχάσω εκ μέρους όλων των εκτελεστικών διευθυντών, των συναδέρφων μου, ότι έχουμε δεσμευτεί απόλυτα για να κάνουμε αυτό που μας έχει ζητηθεί να κάνουμε στα πλαίσια της εντολής μας. Και προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικοί μεταξύ μας υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπέρ των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό είναι κάτι που έχουμε όλοι στο μυαλό μας και στο κεφάλι μας. Τώρα, μετά θα έρθω πιο συγκεκριμένα, ε, γιατί ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, αλλά σε αυτό θα έρθω μετά. Όσον αφορά τη διαφάνεια, για μας η διαφάνεια είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό για σας που είσαστε Επιτροπή Προϋπολογισμών για να μπορείτε να ασκείτε ε, τις δικές σας αρμοδιότητες, ε, να ελέγχετε τα δημοσιονομικά. Αλλά είναι η διαφάνεια εξίσου σημαντική και για τους δικούς μας οργανισμούς, για τον καθένα μας, γιατί αποτελεί βασικό στοιχείο της δημοκρατίας. Το πώς εκτελούμε το έργο μας, τι πόρους έχουμε γι' αυτό και πώς φέρουμε σε πέρα στις αρμοδιότητές μας. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Αυτό είναι κάτι αποδεκτό από όλου. Οπότε όσον αφορά τη διαφάνεια, τη θέλουμε, όπως θέλουμε και την αποτελεσματικότητα, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να συνδυάσουμε κονδύλια με αρμοδιότητες και καθήκοντα που έχουμε. Αυτό είναι κάτι που έτσι κι θέλουμε να το κάνουμε και ελπίζω να το βλέπετε. Αν δεν το βλέπετε είμαστε στη διάθεσή σας ως δίκτυο ή ο κάθε οργανισμός χωριστά. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας δώσουμε ό,τι πληροφορίες θέλετε. Επίση πρέπει να είμαι ξεκάθαρος και για κάτι ακόμα. Όσο περισσότερα καθήκοντα να λαμβάνουμε, χρειαζόμαστε και περισσότερους πόρους για να τα βγάλουμε πέρα. Τώρα, αν εσεί ω νομοθέτης αποφασίσει ότι πρέπει να έχουμε λιγότερα καθήκοντα, εντάξει πάλι, με διαφάνεια, αλλά αυτό σημαίνει λιγότερους πόρους και λιγότερο προσωπικό. Δηλαδή αυτό ισχύει και προ τη μία και προ την άλλη κατεύθυνση. Τώρα, όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών, ήταν κάτι που εμένα με εξέπληξε και πιστεύω και πολλούς από τους διευθυντές μας. Τι, το ότι τελικά διαπιστώνουμε ότι έχουμε πολύ περισσότερα κοινά από ό,τι διαφορετικά στοιχεία μεταξύ μας. Και σας έδωσα ε, κάποια παραδείγματα για τις σχέσεις που είχαμε με τους οργανισμούς που ασχολούνται με τις μεταφορές ή με την υγεία κτλ. Και ο δικός μου ο οργανισμός έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά υπήρχαν δυσκολίες στο θέμα της απολύμανσης και τα λοιπά. Ήταν πράγματα τα οποία τα γνωρίζαμε. Αυτό που δεν είχαμε καταλάβει είναι πόσα κοινά έχουμε μεταξύ μας. Και η κρίση αυτή σε αυτό μας βοήθησε. Για να μπορέσουμε έτσι από κοινού να βρούμε λύσεις στο πρόβλημα. Τώρα, Είμαστε σίγουροι ότι έχουμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο σε όλη τη διαδικασία ανάκαμψης και πάλι προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πολιτών της. Τώρα το ζήτημα που ανέφερα πριν που μένει να σας εξηγήσω και που εμείς ως δίκτυο το κοιτάμε. Κοιτάξτε, εμείς ως οργανισμοί και εσείς ως νομοθέτες δημιουργήσαμε ε, κάποιους ανεξάρτητους οργανισμούς με πόρους που είναι ανεξάρτητοι του ενός από του άλλου. Και είναι κάτι απόλυτα κατανοητό για μας το γιατί έχουν γίνει έτσι τα πράγματα. Όμως αυτό σημαίνει ότι έτσι εμποδίζεται και συνεργασία μεταξύ μας. Είναι ένα εμπόδιο, παρόλο που το εμπόδιο αυτό είναι ένας καλός ε, τρόπος ώστε να δρούμε και οικονομικά. Πάντως, ο λόγος για τον οποίο όσον αφορά ε, τον προπολογισμό δεν είμαι σε θέση να σας δώσω μια κοινή απάντηση για όλους τους οργανισμούς, αλλά θα έπρεπε να διαφοροποιήσω και μπορείτε να απευθυνθείτε στον κάθε οργανισμό χωριστά. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι τα εξή δύο. Πρώτον, ότι συνολικά ο προπολογισμό που έχουμε δει τουλάχιστον μέχρι τώρα για τους διάφορους οργανισμούς δεν σημαίνει ότι πρέπει να μας αφαιρεθούν καθήκοντα. Αυτό σημαίνει ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί τους στόχους της, διατηρεί το επίπεδο φιλοδοξίας της σε σταθερό επίπεδο και τη χρηματοδότηση, αυτό δεν ισχύει μόνο για τους οργανισμούς, για όλα, ενώ απ' την άλλη αν μειωθεί η χρηματοδότηση, αυτό σημαίνει ότι οι οργανισμοί θα μπορούν να κάνουν λιγότερα και θα πρέπει οι μέλη να κάνουν περισσότερα. Οπότε αυτή είναι η εξίσωση. Και εδώ είναι που πρέπει να αναρωτηθούμε πώ μπορούν να ε, γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Ε, τα διάφορα αυτά καθήκοντα μπορούν να γίνουν καλύτερα σε επικουρικότητα με τις χώρες μέλη. Εμείς να το αναλύσουμε και να δούμε. Ή μήπως όχι. Όσον αφορά το περιεχόμενο του έργου μας, για το κλίμα ρωτήσατε, για παράδειγμα, και για την τον οργανισμό περιβάλλοντος. Δεν μπορώ να σα απαντήσω για τον οργανισμό περιβάλλοντος μεν, αλλά όσο δίκτυο εμείς βλέπουμε ότι το έργο του κάθε οργανισμού είναι να συνεισφέρει στην Πράσινη Συμφωνία. Ε, και αυτό το έχουμε υπόψη μας στο πλαίσιο του έργου μας. Έχουμε συζητήσει, έχουμε αναλύσει και μάλιστα ε, στα πλαίσια ομάδων οργανισμών για να δούμε πώς μπορούμε ε, μεταξύ μας να συνεισφέρουμε πιο αποτελεσματικά υπέρ των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, ο δικός μου οργανισμός ε, συμμετέχει στην ίδια ομάδα με τον Οργανισμό για το Περιβάλλον, για την ασφάλεια τροφίμων, για την πρόληψη και έλεγχο νόσων κλπ. Και προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε καλύτερα να ανταποκριθούμε στους πολιτικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους σπόρους, αναφέρθηκα στους σπόρους αρκετά μέχρι τώρα, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα. Εμείς θέλουμε κατάλληλη χρηματοδότηση για τα καθήκοντα που αναλαμβάνουμε. Ο δικός μου οργανισμός, αλλά και άλλοι οργανισμοί για τους οποίους γνωρίζω αρκετά πράγματα, είμαστε περήφανοι για αυτά που έχουμε κάνει. Αλλά μερικές φορές η δουλειά πάει πιο γρήγορα και από τι ίδιε τι πολιτικέ. Οπότε οι πόροι δεν έχουν έρθει ακόμα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούμε, γι' αυτό και ζητάμε ευελιξία. Τέλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θετικά σα σχόλια. Πολύ Χαρικά που ήμουνα και στην Ελεγκτική Επιτροπή όπου το Ελεγκτικό Συνέδριο παρουσίασε τις απόψεις του για τους διάφορους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και είπε ότι γενικά είναι πολύ αποτελεσματική και αποδοτική στο έργο τους προκειμένου να ανταποκριθούν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χαίρομαι που είμαι και εγώ ένας από τους 48 τέτοιους οργανισμούς που παίζει αυτό το θετικό ρόλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρο. ευχαριστούμε πολύ κύριε Χάνσεν και ευχαριστώ βέβαια και όλου του ευρωβουλευτέ που πήραν το λόγο. Οπότε έτσι ολοκληρώσαμε το σημείο 3 στην ημερήσια διάταξη που έχουμε για σήμερα και περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης που είναι η μελέτη για την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εδώ καλωσορίζω πάλι εξ αποστάσεως τον κύριο Νέσμπιτ που είναι από το Ινστιτούτο για τις ευρωπαϊκές πολιτικές για το περιβάλλον, ο οποίος έχει συντάξει μεταξύ άλλων μελέτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Είδαμε πόσο δύσκολο ήταν να φτάσουμε στο 20% για την τρέχουσα περίοδο. Για την περίοδο 2021-2027, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν ως στόχο το 30%. Είναι ρεαλιστικός αυτός ο στόχος, μπορεί να επιτευχθεί και πώς μπορούμε να ξέρουμε τι πρόοδος επιτυχάνεται προς τον στόχο αυτό. Χρειάζεται λοιπόν μία γερή μεθοδολογία. Γι' αυτό λοιπόν και έχουμε σήμερα τον κύριο Νέσπιτ, θα ακούσουμε τι έχει να μας πει και στη συνέχεια εννοείται ότι θα υπάρξουν ερωτήσεις και παρεμβάσεις. Παρακαλώ κύριε Νέσπιτ, έχετε το λόγο για 15 λεπτά. Thank you, Chairman. And... Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ζητώ συγγνώμη που δεν μπορούσα να έρθω και αυτό προσώπως για να σας παρουσιάσω την έκθεση. Δυστυχώς η κυβέρνηση μου αποφάσισε ε, ότι απαιτείται καραντίνα για όσους επιστρέφουν από το Βέλγιο. Θα προσπαθήσω εν συντομία να σας παρουσιάσω την έκθεση. Περνάμε στην πρώτη διαφάνεια που παρουσιάζει γενικά τις αδρές γραμμές της έκθεσης, τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου, τα βασικά τοπορίσματα σε σχέση με το τρέχον ΠΔΠ και τις αρχικές προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Εμείς προτείνουμε να περάσουμε σε ένα νέο, πιο σχολαστικό, πιο εμπεριστατωμένο και αυστηρό μηχανισμό, όπως αναφέρατε και εσείς, κύριε Πρόεδρε. Και επίσης θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για κάποιες εξελίξεις που έλαβα χώρα μετά την οριστικοποίηση της έκθεσης. Γιατί αυτή έγινε πριν α, μετατραπεί σε βασικό παράγοντα διαμόρφωση κατάσταση πανδημία COVID. Επίσης, ε, και για το, την παρακολούθηση της ε, βιοπικιλότητας ε, έχουμε κάποια σύντομα συμπεράσματα, αλλά κυρίως επικεντρωνόμαστε στην παρακολούθηση του κλίματος. Καταρχήν κάνουμε μια γενική επισκόπηση των μεθοδολογιών για την παρακολούθηση του δαπανών στο τρέχον πιδελταπή. Εντοπίζει κάποιες αδυναμίες των προτάσεων και προσπαθούμε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστούν αυτές οι αδυναμίε και πώς θα υλοποιηθεί ο στόχος του 25%. Επίσης, είμαστε υπέρ ενό πιο αυστηρού συστήματος. Θέλουμε φυσικά να βοηθήσουμε την Επιτροπή στο έργο για το επόμενο ΠΔΠ. Ε, μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου εκπονήσαμε την έκθεση. Το αρχικό της σχέδιο υπευλήθη στις αρχές Μαρτίου, οπότε δεν λάβαμε υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις της πανδημίας COVID και τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δαπάνες ε, του σχεδίου ανάκαμψης του Next Generation EU. Ποια είναι τα βασικά μας πορίσματα για το τρέχον ΠΔΠ. Το βασικό στοιχείο είναι ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν παρακολουθεί τις δαπάνες για το κλίμα, δηλαδή ε, δαπάνες που πρωταρχικός του στόχος είναι ε, οι κλιματικοί στόχοι, αλλά ε, οι δαπάνες που συμβάλλουν στους κλιματικούς στόχους. Οπότε μπορούν να αναφέρονται σε άλλα θέματα, οικονομική ανάπτυξη, εδαφική συνοχή, οι ε, αγροτικές, ε, αγροτικά εισοδήματα. Επίσης, έχουμε διαφορετική προσέγγιση από τον ΩΣΑ, γιατί εκεί αναφέρεται πρωτοχικός ή μείζον στόχος της δαπάνες αντί να εξετάζει το κατά πόσο οι δαπάνε ε, συμβάλλουν κατά μείζωνα τρόπο ή μετρίωση στην συνεισφορά των, ε, στην, ε, συμβάλλουν στους κλιματικούς στόχους. Και επίσης η βιοπικιλότητα δεν εντάσσεται στη παρακολούθηση που κάνει όσα. Ένα άλλο θέμα που παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει κάποιος γενικός οριζόντιος μηχανισμός είτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε στα άλλα θεσμικά όργανα ώστε να κατανείμονται τα κονδύλια για την υλοποίηση του στόχου του 20%. Δεν υπάρχει αντίστοιχος μηχανισμός για να μειώνονται ε, οι δαπάνε σε ένα τομέα όταν αυξάνονται σε άλλον. Επίσης, έχω μια τάση να επικρίνουμε μηχανισμούς παρακολούθησης, ιχνηλάτησης, αλλά ε, είναι πρωτοφανή αυτός ο μηχανισμός, αν προηγουμένου δεν υπάρχουν αντίστοιχοι εθνικοί μηχανισμοί για να μπορέσουμε να το συγκρίνουμε με κάτι άλλο. Και παρά τις αδυναμίες του, είναι αρκετά σημαντική αυτή η μεθοδολογία. Και απαράμιλη. Τώρα, βασικά πορίσματα. Ε, βασικά προγράμματα που συμβάλλουν στο στόχο του 20% είναι η κοινή γεωργική πολιτική και η πολιτική συνοχή. Δηλαδή το Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και Περιφερειακή Ανάπτυξη και από την πολιτική συνοχή το Ταμείο Περιφερειακή Ανάπτυξη και το Ταμείο Συνοχή. Η προσέγγιση του πρώτου πυλώνα ε, με το Ταμείο Εγγυήσεων, το Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων της ΚΑΠ, ακολουθεί την εικασία ότι τρεις προϋποθέσεις ε, του πρασινίσματος των άμεσων ενισχύσεων που έχει τρία, σκέλη, δηλαδή την προϋπόθεση των μόνιμων υποσκοτόπων, που θεωρεί, θεωρείται ότι συμβάλλει κατά 100% στους οικολογικούς στόχους. Κατά 40% ε, συμβάλλουν οι περιοχές οικολογικής εστίασης, ενώ η διαφοροποίηση των καλλιεργιών ε, θεωρείται ότι δεν συμβάλλει στην υλοποίηση των κλιματικών στόχων. Επίσης, υποθέτει το 1 πέμπτο του υπόλοιπων ε, άμεσων ενισχύσεων συμβάλλουν με τρίος, κατά 40%. Επικρίθηκε αυτή η προσέγγιση από το ελεκτικό συνέδριο του 2016 ως υπερβολικά γενναιόδορη και οδηγεί σε 19,46% του υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων. Επίσης, ε, το Γεωργικό Ταμείο Περιφερειακής ε, Αγροτικής Ανάπτυξης ε, στηρίζει κυρίως στις εστιασμένες περιοχές και υπολογίζει κατά 100% τα, τα κλιματικά αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και μια μετάβαση προς οικονομία χαμηλού άνθρακα. Επίσης, 40% χρησιμοποιούνται κάποια μέτρα για την αποφύγη του κινδύνου στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Οι δαπάνε της ε, συνοχής στηρίζονται στη, σε κάποια τομείς παρέμβασης που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των προγραμμάτων δαπανών. 100% είναι ο δείκτης ε, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 40% για άλλους ε, τομείς. 100% είναι για την ανανεώσιμη ενέργεια, για την ενεργειακή αποδοτικότητα και ο δείκτης του 40% εφαρμόζεται σε παρεμβάσεις στους σιδηροδρόμους, τους θαλάσσιους λιμένες, πολυτροπικές μεταφορές και ούτω καθεξής. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες για το φάσμα των άλλων κονδυλίων, Πάντως, ε, το, ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλίας έχει κάποια μέτρα που ε, έχουν το δίκτυο 100% όπως η μόνιμη πάυση των αλευτικών δραστηριοτήτων. Ή έχουμε άλλα μέτρα ε, όπως το ορίζοντας 2020 που συμβάλλουν στο μετριασμό των κλιματικών αλλαγών, όπως η μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλή χρήση άνθρακα, αλλά και το πρόγραμμα LIFE συμβάλλει. Και έχουμε κάποιε δημοσιονομικέ γραμμέ ε, εξωτερικών δαπανών που επίση συμβάλλουν, κυρίω η αναπτυξιακή βοήθεια. Περνάμε τώρα στην επόμενη διαφάνεια. Όπως είπα, το σύστημα είναι ίσως και το πιο αναπτυγμένο στις, ε, το πιο προηγμένο στις αναπτυγμένες χώρες. Έχει κάποια πλανεκτήματα, όπως χαμηλό μικρό διοικητικό ε, και προσπαθεί να αξιοποιήσει κάποια παράλληλα ωφελήματα. Έχει όμως και αρκετές αδυναμίες. Για παράδειγμα, είναι κατά προσέγγιση. Δεν στηρίζεται σε μια λεπτομεριακή σχολαστική και περιστατωμένη προσέγγιση της παρακολούθησης. Γι' αυτό φυσικά έχει και μικρό διοικητικό άχθος. Επίσης, σε κάποιους τομείς, όπως στην κοινή γεωρική πολιτική και στο Ταμείο Θάλασσας και ε, υπάρχει υπερβολικά γενναιόδορη ευνοϊκή μεταχείριση. Ούτε απαιτεί από τα προγράμματα να επιδείξουν ε, αποτελέσματα και να αποδείξουν την υλοποίηση των στόχων. Επίσης, ε, δεν αντιμετωπίζει τους κινδύνους στο αρνη, τους αρνητικούς για το κλίμα. Και επίσης δεν κάνει διάκριση μεταξύ των δαπανών για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές είναι πολύ δύσκολο να χρησιμοποιηθεί ο μηχανισμός χνηλάτιση παρακολούθησης για να διαφοροποιηθούν τα κονδύλια που αφορούν το μετριασμό από τα κονδύλια που αφορούν το, την προσαρμογή. Επίσης, δεν συνδέεται επαρκώς στην πολιτική διαδικασία για τη συμφωνία του ετήσιου προϋπολογισμού. Για το επόμενο τώρα, Δελταπή, Η πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά υιοθετεί την ίδια προσέγγιση με το τρέχον πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουμε κάποιε βελτιώσει, κυρίω το γεγονό ότι έχουμε μία των προτέρων εξάντε προσέγγιση για την αξιολόγηση του τρόπου υλοποίηση του στόχου του 25% και επίση ε, προσπαθεί να εξασφαλίσει παρόμοια είδη σχεδίων σε διαφορετικά προγράμματα να αξιολογούνται με τον ίδιο τρόπο. Είναι πιο συνεκτικός ο τρόπο και η προσέγγιση που χρησιμοποιεί στο επόμενο ΒΔΠ. Κάποιες αλλαγές έγιναν στη χρήση των δικτών 40 και 100%. Υπάρχουν κάποιες αλλαγέ, ε, ώστε ε, να λαμβάνονται περισσότερες λεπτομέρειες στους τομείς παρέμβασης και επίσης ε, τα μέτρα για τις επενδύσεις στους σιδηροδρόμους πέρασαν από το δίκτυο του 40% στο δίκτυο του 100%. Επίσης, ε, μια πιο αυστηρή προσέγγιση οθετήθηκε για τις περιοχές ε, με φυσικούς περιορισμούς. Υιοθετεί πιο επιφυλακτική προσέγγιση και υπολογίζεται με το δίκτυο του 40% και όχι το 100%. Βέβαια, το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι έχει πολύ πιο γενναιόδορη προσέγγιση για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο ε, Εγγυήσεων. ίσως δεν είναι Ευανάγνωστο ο πίνακας και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Πάντως η κάτω γραμμή του πίνακα δείχνει ότι αν οι δαπάνες, πληρωμές για τις δαπάνες είχαν χρησιμοποιούνταν με βάση το προηγούμενο πι που κρίθηκαν από το ελεκτικό συνέδριο στις υπερβολικά γενναιόδορες θα, συνέβαλαν, θα συνέβαλαν κατά 4,6% μόνο στο, στο συνολικό προϋπολογισμό για το κλίμα. Το συνολικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και όχι μόνο το προϋπολογισμό του Γεωργικού Ταμείου Επενδύσεων. Οπότε θα χρειαστούν περισσότερες ε, επενδύσεις από τα κράτη-μέλη για τα οικολογικά συστήματα. Αλλά το πολύ πολύ να φτάσουμε στο 52% σχέση με τον συνολικό στόχο, δηλαδή 12,26% του συνολικού ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Οπότε έχουμε 7,5% αύξηση από τις αλλαγές στον υπολογισμό του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για τις επενδύσεις, για τις ε, εγγύησεις, συγγνώμη. Και έτσι αν έχουμε αύξηση του κλιματικού στόχου από 20-25% θα έχουμε δυσκολία γιατί μόνο το 7% θα υλοποιήσουμε και αν θέλουμε από το 25% να περάσουμε στο 30% η κατάσταση θα είναι ακόμη πιο δύσκολη. Όπως είπα και προηγουμένως, είτε θα πρέπει οι συνομοθέτες να αυξήσουν ριζικά τις κλιματικές φιλοδοξίες στην πρόταση του πιδελταπή είτε θα πρέπει να υιοθετήσουν μια πιο συντηρητική προσέγγιση της παρακολούθησης για το Γεωργικό Ταμείο, Κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να περιθεί μεγαλύτερη ε, περιβαλλοντική προσέγγιση από άλλα προγράμματα για να υλοποιηθεί ο στόχος του 25% και του 30% που είναι η νέα φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σε ό,τι αφορά το γενικό σύστημα υποβάλαμε διάφορες προτάσεις, την ανάγκη για σαφείς πολιτικές αποφάσεις για τη μεθοδολογία του κάθε προγράμματος ό,τι αφορά τον υπολογισμό των κλιματικών δαπανών, σαφή διάκριση μεταξύ των ε, δαπανών για το μετριασμό των κλιματικών αλλαγών και των δαπανών για την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης, να περιλαμβάνονται μόνο προγράμματα που έχουν ε, ε και κατά προτίμηση ποσοτικοποιημένους κλιματικούς στόχους και μάλιστα σε ένα αρκετά απαιτητικό επίπεδο. Να αναφέρονται για παράδειγμα τόνοι διοξιδίου του άνθρακα που εξοικονομούνται ανά ευρώ. Επίσης, θέλουμε ενισχυμένους μηχανισμούς για να αποφευθούν ε, αρνητικοί αντίκτυποι στο κλίμα ή τη βιοπικιλότητα και να, συνδεθεί καλύτερα, ε, να συνδεθούν καλύτερα οι κλιματικές δαπάνες με τα εθνικά ε, σχέδια ενέργειας και κλίματος. Το προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά θέλαμε μια μεγαλύτερη αυστηρότητα. Θα είναι βέβαια πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο από την αρχή του επόμενου ΠΔΕΛΤΑΠΗ, αλλά θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει την εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων και να εισαγάγει σταδιακά το νέο σύστημα. Επίσης, πρόσφατες εξελίξεις. Η αρχική στόχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούσε το 25%. Το, η μετάβαση από το 25% στο 30% θα κάνει πολύ πιο δύσκολη την ε, εφαρμογή, ιδιαίτερα αν, μια, αν, δεν, αν δεν λάβουμε μια πιο συντηρητική προσέγγιση στις αγροτικές δαπάνες. Και η καθυστέρηση της συμφωνία του ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ καθιστά ακόμη πιο δύσκολη την υλοποίηση του 30%. Αν μείνει το Ταμείο Εγγυήσεων στο 19, γύρω στο 20%, αντί για 50% για ένα μόνο χρόνο, θα έχουμε περίπου 1% του συνολικού ΠΙΔΕΛΤΑΠΗ που θα πρέπει να προέλθει από αυξημένη ε, κλιματική συμμετοχή άλλων προγραμμάτων. Και αν συνεχιστεί αυτό ακόμη ε, για, ένα δεύτερο, μια δεύτερη χρονιά, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο το χάσμα. Επίσης, ε, αν αναγνωρίσουμε ότι η καθυστέρηση στην εισαγωγή των νέων ρυθμίσεων για την ΚΑΠ θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη αύξηση του χάσματος, θα πρέπει να έχουμε μια ριζική ε, επανεστίαση των προτεραιοτήτων για την επιμερισμένη διαχείριση ώστε να ληφθεί υπόψη το κλίμα. Θα χρειαστεί μια πιο συντηρητική προσέγγιση στις δαπάνες της ΚΑΠ. Σε ό,τι αφορά τι ε, δαπάνες του νέου σχεδίου ανάκαμψη, του Next Generation EU, Δυστυχώ δεν έχουμε μηχανισμούς που να περιλαμβάνονται στην νομοθετική πρόταση για να υλοποιηθεί αυτή η παρακολούθηση, αυτή η χνηλάτη, στο tracking. Και νομίζω ότι περισσότερο στηριζόμαστε σε ευσεβείς πόθους και υπερβολικές εκτιμήσεις και όχι στην πραγματικότητα. Επίσης, ε, ε, ο μηχανισμός για την αθεκτικότητα έχει ακόμη πιο αυστηρή προσέγγιση για το, την παρακολούθηση ό,τι αφορά το κλίμα. Γι' αυτό καλό θα ήταν αυτός ο μηχανισμός, αυτή η διευκόλυνση για την αθεκτικότητα να έχει αντίστοιχο μηχανισμό παρακολούθησης. για να φανεί ποια θα είναι η συμβολή του κλίματος σε αυτές τις δαπάνες. Αυτό θα έπρεπε να είχαν ζητήσει οι συνομοθέτες. Αυτά εν συντομία κύριε Πρόεδρε, μια πολύ σύντομη επισκόπηση ε, των αδρόγραμμών της έκθεσής μας και πολύ ευχαριστώ ε, να απαντήσουμε στις απορίες σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Νέσβητη για την παρουσίαση αυτή και που τηρήσατε σε μεγάλο βαθμό το χρόνο. Πάμε στους ομιλητές ε, και πρώτα απ' όλα στους τρεις ευρωβουλευτές ε, που ήταν επιφορτισμένοι με την παρακολούθηση αυτής της μελέτης. Πρώτα απ' όλα η κυρία Γκουαρδία Ζαμπάλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για την πρόταση και για τις ε, επεξηγήσεις όσον αφορά τη μελέτη αυτή. Μιλάω και εκ μέρου τη κυρία Μάρκες, η οποία ήταν σε κάποια άλλη, ε, σε κάποια άλλη συνεδρία, έχουν καθυστερήσει και γι' αυτό δεν μπορεί να είναι εδώ, μου έχει δώσει ένα σημείωμα. Η κλιματική αλλαγή ήταν το κύριο θέμα στις εκλογέ, στι ευρωεκλογέ που είχαμε το 2019 σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο, όχι μόνο οι νέοι, αλλά όλοι ενδιαφέρονται πολύ για τον, πολίτη, για τον πλανήτη και για το περιβάλλον. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να αποκριθεί στους Ευρωπαίους πολίτες ε, όσον αφορά τις ανησυχίες τους και τόσα εμείς ε, βάλαμε στα θέματα στις ευρωεκλογές και πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολιτικές μας την κλιματική αλλαγή. Οι διάφορες τέτοιες πολιτικές χαρακτηρίζουν το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και σε αυτή την περίοδο και πρέπει να το κάνουν ακόμα περισσότερο για την περίοδο 2021-2027. Συνεπώς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το νέο αυτό Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τον Οκτώβριο που μας πέρασε, ζήτησε ένα ποιοτικό άλμα όσον αφορά τις πολιτικές προσπάθειες και τις οικονομικές προσπάθειες της Ευρώπης για να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή σε όλες τις πολιτικές. Οπότε έχουμε βάλει δίκτυ όσον αφορά τις δαπάνες μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αυτό είναι το 30%. Αυτό σημαίνει ότι ο προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για να επιτευχθούν οι πολιτικέ αυτέ κατά τη κλιματική αλλαγή. Όμω, ω αρχή που είμαστε για τον προπολογισμό, χρειαζόμαστε μια μεθοδολογία οποία να είναι αποτελεσματική, με διαφάνεια, για να παρακολουθήσουμε τι δαπάνε και το επίπεδό του, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό το 30%. Και γι' αυτό και ζητήσαμε τη μελέτη αυτή από τους εμπειρογνώμονες για να τους ακούσουμε και να δούμε πώς θα συμπεριληφθεί καλύτερα το περιβάλλον στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό. Ο κύριος Νέτβικ μελέτησε τις σημερινές μεθοδολογίες όσον αφορά τις δαπάνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα. Αυτός ήταν ο στόχος της μελέτης αυτής εξάλλου. Συνεπώς, είναι ένα πρώτο μικρό βήμα που κάνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση και το λέω και το λέει και η κυρία Μάρκες γιατί χρειαζόμαστε αλλαγές στη μεθοδολογία στις ε, πολιτεις δημοσιονομικες δημοσιονομικές προοπτικές 2021-2027 και ένα νέο μηχανισμό παρακολούθησης που να είναι πιο αποτελεσματικός. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το κάνει και να φροντίσει να επιτευχθεί αυτό για το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο κύριο Νέσκερ μα έδωσε κάποια στοιχεία για το τι θα πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε αυτό το 30% στο επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Όμω, μια που δεν είχε αρκετό χρόνο, ίσω θα μπορούσε να επικεντρωθεί στις συμβουλές του αυτές ακόμα περισσότερο για να μας πει πώς μπορούμε να έχουμε μια νέα πιο αποτελεσματική μεθοδολογία και περισσότερη διαφάνεια ώστε να πετύχουμε αυτό το 30% που ζητούμε όσον αφορά τις δαπάνες μας σε σχέση με το κλίμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σχόσνικ από το when we came out with this with this study. Uh, oh, no, thank you. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Νέσμπιτ και αγαπητοί συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Πολύ καλή στιγμή γιατί αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο Όλη η παρουσίαση εστιάζεται στις δαπάνες για το κλίμα και χαίρομαι που καλύπτονται εν μέρη χωρίς παραπάνω δαπάνες γιατί δεν έχουμε μόνο το κλίμα ως πρόβλημα. Έχουμε και τη βιοπικιλότητα, οπότε πρέπει να τα εξετάζουμε και τα δύο. Και χαίρομαι που ζητήσαμε 10% στόχο δαπανών εδώ για τη βιοπικιλότητα. Τώρα η μελέτη δεν θα αποτελέσει λύση για τα πάντα παρότι είναι πολύ ωραία. Αλλά δεν είναι παρά μία απόπειρα. Δεν είναι η μόλι μελέτη. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη μελέτη του ελεγκτικού συνεδρίου, που είναι πολύ σημαντική για την ε, συζήτηση αυτή. Να έχουμε το καλύτερο σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγματι, αν το κοιτάξουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι τέλειο. Απλά είναι καλύτερο από τα άλλα. Και αυτό μας προκαλεί να γίνουμε καλύτεροι, να βελτιωθούμε, να βελτιώσουμε τον τρόπο επίτευξης των στόχων για το κλίμα. Κάτι άλλο που θέλω να θίξω είναι το γεγονός ότι δεν είναι όλα τα προβλήματα εξίσου σημαντικά. Τόσο για το κλίμα όσο και για τη βιοπικιλότητα. Όπως για παράδειγμα ο προπολογισμό ε, για την αμυντική συνεργασία είναι κατά την απόψη μου λιγότερο σημαντικός. Οπότε δεν πρέπει να, κάνουμε, να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα με τον ίδιο τρόπο, να εξετάζουμε πρόγραμμα προς πρόγραμμα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε τη λογιστική και τους υπολογισμούς σωστά, ανάλογα με τους στόχους. Και για να επιτευχθεί το συνολικό 30% και το 10% και οι δύο αυτοί στόχοι. Οπότε να μην μένουμε σε κενά λόγια, πρέπει να δράσουμε. Οπότε αναμένω να συνεργαστούμε και με τον σκιώδη για την ταξονομία, που πιστεύω ότι είναι μια νομοθεσία που θα μας βοηθήσει για να κάνουμε τους λογιστικούς υπολογισμού σωστά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για τους ε, πρασίνους, ο κύριος Αντρέσεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστούμε κύριε Νέσπιτ για την μελέτη και για την παρουσίαση σήμερα. Πιστεύω ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Κατάλληλη στιγμή διότι αυτή τη στιγμή διαπραγματευόμαστε το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και τον ετήσιο προπολογισμό με στις επόμενες εβδομάδες καθώς και άλλα στοιχεία όπως την κλιματική νομοθεσία, την πρώτη ευρωπαϊκή κλιματική νομοθεσία. Οπότε τώρα πρέπει να τα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Και πολλά είναι τα ζητήματα που τίθενται όσον αφορά όλα αυτά τα θέματα. Το γεωργικό κομμάτι φυσικά είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα. Επίσης ε, το κλίμα, ε, συγγνώμη γεωργία πόσο συνεισφέρει στο κλίμα, ουσιαστικά και άλλα στοιχεία, αλλά θα ήθελα να εστιαστώ σε δύο πράγματα, για τα οποία θα ήθελα να μάθω λίγα παραπάνω. Ποια είναι η δική σας άποψη κύριε Νέσπιτ, διότι πιστεύω πραγματικά ότι θα παίξουν ρόλο κλειδί για να έχουμε έναν αποτελεσματικό προπολογισμό μέσα στα επόμενα έτη. Η μελέτη σας δείχνει ότι υπάρχουν πολλά παραθυράκια και κενά στον τρόπο με τον οποίο υπολογίζουμε ε, τις ε, ευθύνες και το μερίδιο του κλίματος στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. Και όπως υπόθηκε ήδη, πρέπει να γίνουν πολλές προσπάθειες βελτίωσης. Οπότε θα ήθελα να σας ρωτήσω, ε, η αρχή αυτή του να μην βλάπτεις, do no harm, υπάρχουν πολλά συγκεκριμένα μέτρα που σχετίζονται με τον ευρωπαϊκό προπολογισμό και τα οποία θεωρούμε προβληματικά, διότι κάποια έργα ζημιώνουν το περιβάλλον. Αυτό πρέπει λοιπόν να αλλάξει. Είχαμε αποφασίσει ένα ψήφισμα για το σε νομικό πλαίσιο, ώστε να περιλαμβάνει την αρχή ε, του να μην βλάπτεις ε, do no harm στο επόμενο κανονισμό για... είναι και κομμάτι των συμπερασμάτων του Συμβουλίου και τώρα θα πρέπει να κάνουμε πιο συγκεκριμένα βήματα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω, έχετε πιο συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς μπορεί να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτής της αρχής ε, του να μην βλάπτεις, όπως για παράδειγμα το να αποκλείονται διάφορα ε, έργα ή άλλα στοιχεία. Ή έχετε άλλες συστάσεις θα ήθελα να μάθω περισσότερα. Και το άλλο ζήτημα αφορά του στόχους βιοπικιλότητα. Το ανέφερε ήδη ο κύριος Χόισεκ. Προτείνουμε στόχο 10% για τη βιοπικιλότητα όσον αφορά το πολιτισμό στο νομικό πλαίσιο. Αυτό που θα ήθελα να μάθω από εσά ποιε είναι οι απόψεις όσον αφορά την εξέλιξη του στόχου βιοποικιλότητας και του μεθοδολογίας παρακολούθησης. Θα πρέπει να μοιάζει με αυτό που κάνουμε για το κλίμα ή πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό. Τόσο η στοχη όσο και η μεθοδολογία μεταξύ βιοποικιλότητας και κλίματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από τους άλλους ομιλητές υπάρχει κάποιο από το ΕΛΚΑ, ο οποίο θα ήθελε το λόγο. Κυρία Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έχω μια παρατήρηση και οι δύο κύριοι μίλησαν για μια πολιτική με στόχους. Ε, η κυρία Μπέργκερ είχε μιλήσει για αυτόν τον τομέα, μια υπηρεγνώμων που γνωρίζουμε και εκτός της ε, Αυστρίας. Ε, έχετε... Δεν την έχετε ρωτήσει από την ομάδα σας και αυτό μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ευχαριστούμε κυρία Λαπόρτ. ID. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η μελέτη αναλύει αντικειμενικά την κατάσταση και εξετάζει τη μεθοδολογία για το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η δράση για το κλίμα θα βρίσκεται στο επίκεντρο με τεράστια ποσά. Πρέπει λοιπόν η μεθοδολογία να είναι πιο διαφανής και πιο ακριβής από ό,τι παλιότερα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τον Νοέμβριο του 2018 είχε προτείνει η παρακολούθηση να γίνεται βάση δικτών απόδοσης νέων με διάκριση μεταξύ μετριασμού και προσαρμογής. Η προηγούμενη Επιτροπή ήθελε 25% του ευρωπαϊκού προπολογισμού να αφιερώνεται στο κλίμα για το επόμενο διάστημα μεταξύ 2021 και 2027 σε αντίθεση με το 20% που έχουμε για την τρέχουσα περίοδο, 14 με 20. Και θέλουμε να πρέπει στο 30% στο επόμενο σε δημοσιονομικό πλαίσιο αυτός ο αριθμό Δεν θα μειωθεί αυτό ο αριθμό ε, λόγω της πανδημίας του, ε, του κορονοϊού και δεν είναι πολύ ε, αισιόδοξη. Τώρα η Κομισιόν εστιάζεται στους στόχους του κλίματος, στον ενιαίο στόχο της, του κλιματικού μετριασμού και διάφορε δαπάνε για την συνεργασία και την ανάπτυξη. Η μέθοδο που προβλέπεται στην εκθέση αυτή αξιολογεί την νομοθεσία και τα επίσημα έγγραφα για την παρακολούθηση τη δράση για το κλίμα, περιλαμβάνει στόχου συγκεκριμένου και επαληθεύσιμου. Αυτοί οι στόχοι θα αναθεωρηθούν. Επιπλέον, συμφωνώ με τις συστάσεις ε, για τις δαπάνες ε, για το κλίμα να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ προσαρμογής και μετριασμού να υπάρχει σαφή διάκριση μεταξύ τη παρακολούθηση του κλίματο και τη βιοπικιλότητα και των εθνικών στρατηγικών και στόχοι πιο πιστευτοί ε, μεταξύ αυτών που ορίζει η Κομισιόν. Επίση, πρέπει να αναρωτηθούμε ο ρυθμό ε, απαλλαγή από τι ανθρακούχε εκπομπέ. Ο στόχο για το 2030 πρέπει να οριστεί βάσει των αποτελεσμάτων που θα έχουμε στο μέλλον. Η αλλαγή αυτή μεθόδου δεν μπορεί να εφαρμοστεί από το επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο η πράσινη αυτή μετάβαση μέσα στο επόμενο πολιτικο δημοσιονομικό πλαίσιο θεωρούμε ότι πρέπει να προσαρμοστεί στη σημερινή πανδημία και στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σήμερα. Ευχαριστούμε. Κάποιο από το ECR θα ήθελε να πάρει το λόγο, κύριε Τζόνσον. Ε, Σας ευχαριστώ. Πολύ ε, σύντομα. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε τη σοβαρότητα της κατάστασης στο κλίμα αλλά θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και προσεκτικοί κατά τη διατύπωση των στόχων, των κλιματικών μας στόχων. Γιατί έχουμε αυτά τα, τους πράσινους αριθμούς, όπως λέμε, και υπάρχουν πολλές εκτιμήσεις γιατί, και διάσταση απόψεων για το κατά πόσο είναι σκόπιμο όλα αυτά τα νούμερα, τα πράσινα. Επίσης, έχουμε μια σωρία προκλήσεων λόγω της πανδημίας COVID. Και νομίζω ότι το θέμα του κλίματος, αν επικεντρωθούμε μόνο σε αυτό, δεν θα ε, τύχει θετικής ε, υποδοχής ε, στο σύνολο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Γιατί προέχει να αντιμετωπίσουμε την πανδημία COVID. Μερικές χώρες εξαιτίας οικονομικής κρίσης δεν θα έχουν καν δυνατότητα ανάπτυξης δεν θα πρέπει να περιοριστούμε σε δηλώσεις για την ε, εμπιστευτικότητα ή τον απόρριτο χαρακτήρα κάποιων ε, εγγράφων, γιατί τέτοιες δηλώσεις ε, διαταράσσουν τη συζήτηση για το κατά πόσο είναι σκόπιμη όλη η στόχη της, πολιτι... της κλιματικής πολιτικής. Φυσικά θέλουμε να διαφυλάξουμε το κλίμα και το περιβάλλον, αλλά αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ, πολλά άλλα σοβαρά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε πέραν της ε, περιβαλλοντικής πολιτικής και αυτά είδα θα πρέπει να τα μελήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κόκαλης τώρα εκ μέρους της ΓΚΟΕ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ε, πραγματικά σοκάρι. Επιτρέψτε μου να τα πω ομά. Η περιγραφή της κατάστασης πραγμάτων δείχνει ότι δεν έχουμε ένα καλό και σωστό σύστημα, διότι δημιουργεί προβλήματα και προσφέρει μόνο μια επίφαση για πρασίνισμα. Η συνεισφορά αυτή του 30%, του 25% συγγνώμη, σημαίνει ότι το 75% δεν πηγαίνει για το κλίμα και για το περιβάλλον. Και αυτό είναι ακριβώς που σοκάρει με τα, τις προσπάθειες που κάνουμε εξάντε. Εσείς πολύ σωστά βέβαια λέτε και με πολύ θάρρος θα έλεγα μάλιστα ότι η γενική εντύπωση του κοινού που μας εξέλεξε είναι ότι 25% του προπολογισμού θα πάει στο στόχο του κλίματος. Ενώ δεν ισχύει αυτό. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και απέναντι στον κόσμο και απέναντι στους πολιτικούς. Και εμείς αυτό το καταλαβαίνουμε. Συνεπώς, προτείνω εμείς ως Επιτροπή Προϋπολογισμών να σας επιτρέψουμε να συνεχίσετε το έργο σας για να εξετάσετε τις διάφορες γραμμές του προϋπολογισμού για τον επόμενο προϋπολογισμό και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Και πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα και να βασιζόμαστε στην επιστήμη και να διασφαλίσουμε ότι θα φέρουμε σε πέρα όσα μας ζήτησαν οι Στηρίζω λοιπόν τις ιδέες σας και για την ταξινόμηση και για το ου βλάψης και θα ήθελα να ζητήσω από όλους τους συναδέρφους να αγωνιστούν για να έχουμε μια αποτελεσματική μεταρρύθμιση γρήγορα όσον αφορά το σύστημα μέτρησης δεν είναι ένα σύστημα που μπορούμε να υποστηρίξουμε και ούτε θα μας δώσει τα αποτελέσματα τα οποία θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Λαρουτουρού. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Νάσπη για την μελέτη αυτή που είναι τόσο πλήρης αλλά και τόσο ανησυχητική όπως λένε και οι συνάδελφοι. Η κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός. Βλέπουμε τις πυρκαγιές ε, στα δάση, βλέπουμε τους κυκλώνες, 200 ε, χιλιόμετρα την ώρα, είναι πολύ ανησυχητικά όλα αυτά. Βλέπουμε το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Ε, παρά την οικονομική κρίση, σε ένα χρόνο 2,6 μονάδες αυξήθηκε το διοξίδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, περισσότερο από ποτέ τα τελευταία 50 χρόνια. Οπότε κινδυνεύουμε κι εμείς και οι τα κτλ. Δεν μπορούμε να δεχτούμε λοιπόν η δράση της Ευρώπης να οδηγείται από κάτι το ασαφές. Πρέπει να έχουμε δείκτες που θα βελτιωθούν και να βελτιώνονται όχι μόνο ε, με έναν κανονισμό χωρί να έχουμε αλλάξει την ουσία. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν για αυτή τη μελέτη που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, έρχεται για την κατάλληλη στιγμή όπω είπα και οι συνάδελφοι. Δεν θα κερδίσουμε τη μάχη του κλίματο αν δεν έχουμε σωστή πρικοδότηση, σωστό προπολογισμό και σαφεί δείκτε που να είναι κατανοητοί και να υπάρχει και διαφάνεια για αυτού. Όλοι οι συνάδελφοι εδώ στην Επιτροπή Προπολογισμών θέλουν να ξέρουν που πηγαίνει το κάθε ευρώ, πόσο μάλλον για το κλίμα. Τρει ερωτήσει εκ μέρου τη ομάδα μου. Πρώτον, τι συμπεράσματα θα βγάλουν από την μελέτη αυτή, με τι χρονοδιάγραμμα και τι διαδικασία ε, μπορούν να ακολουθήσουν η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο για να έχουν νέους δείκτες πιο αποτελεσματικούς που πρέπει να είναι η κοινή μας προτεραιότητα. Πολύ γρήγορα πρέπει να έχουμε τέτοιους νέους δείκτες. Δεύτερον, πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια από το New Generation EU και τι ε, μαθήματα παίρνουμε από τη μελέτη αυτή. Και κύριε Νέσπιρ, θέλω να ρωτήσω και εσά κάτι. Ανά πρόγραμμα, τι δείκτες προτείνετε, όπως είπε και συνάδελφος ε, από το Ρινιού. Θέλουμε δείκτες που να μιλάνε ε, στον κόσμο, στους αγρότες, στις επιχειρήσεις επιτόπου. Δηλαδή, τι λύπασμα, τι συγκεκριμένα στοιχεία για τον καθένα. Γιατί μόνο αν έχουμε απλούς ε, δείκτες και καλούς δείκτες θα βοηθήσουμε. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, τα επαγγελματικά ατυχήματα μειώθηκαν στα τέσσερα τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε ένα σαφή δείκτη που είναι κάθε χρόνο τι ατυχήματα έχουμε σε κάθε επιχείρηση σε σχέση με το μέσο όρο του κλάδου. Και έχουμε βάλει ένα μπόνους μάλους, οπότε αν μια επιχείρηση έχει παραπάνω από το μέσο όρο πληρώνει περισσότερα, αν έχει λιγότερα ατυχήματα από το μέσο όρο του κλάδου πληρώνει λιγότερα είναι κάτι σαφές, όλοι το καταλαβαίνουν, είναι κάτι που μετριέται εύκολα, επαληθεύεται εύκολα και βοηθάει και τον κόσμο να δράσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αναπρόγραμμα λοιπόν πρέπει να καταλήξουμε σε απλούς δείκτες που να βοηθήσουν τους διάφορου παίκτες του παιχνιδιού να αλλάξουν συμπεριφορά. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Κύριε Νέσβιτ, έχετε το λόγο για να απαντήσετε αν θέλετε. Ε, δέκα λεπτά έχετε στη διάθεσή σας εσείς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τα μέλη που παρενέβησαν. Χαίρομαι για την προσοχή που έχει προσελκύσει η έκθεση αυτή. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη αν δεν κατάφερα να καταλάβω ακριβώς ποιος ε, βουλευτής μίλησε για ποιο θέμα. Για την κυρία Κουέντε Σαβάλ. Αυτό που ανέφερε για τη σπουδαιότητα της κλιματικής αλλαγής ε, στις ε, πρόσφατες ε, ευρωεκλογέ. είναι πολύ σημαντικό. Είναι εύκολο να επικρίνει κανείς το σημερινό σύστημα ως ε, όχι αρκετά αυστηρό στη γενική του προσέγγιση για κάποια προγράμματα. Ωστόσο, η πολιτική οδός που, πρέπει, που ακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι πιο εστιασμένη στην παρακολούθηση του κλίματος. Οπότε οι νομοθέτες διασφαλίζουν και πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι μηχανισμοί που θα χρησιμοποιηθούν για τον στόχο του 30% για τις δαπάνες θα πρέπει να γίνουν ε, λαμβάνοντα υπόψη του Ευρωπαίου πολίτε που ψήφισαν υπέρ τη κλιματική αλλαγή ω σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα ζήτημα για τι ε, γεωργικέ δαπάνε ε, και για κάποιου από του άλλου μηχανισμού που επικρίνει και το ελεγκτικό συνέδριο. Παρομοίω, κάποια μέλη ανέφεραν ότι το σημερινό σύστημα είναι ανεπαρκές. Πιστεύω παρομοίω ότι βρισκόμαστε σε μια φάση εξέλιξη προ ένα πιο αποτελεσματικό ε, σύστημα παρακολούθηση του κλίματο. Αναπόφευκτα, όταν υπάρχει ένα σύστημα και οι θύνοντε, αυτοί που λαμβάνουν τι αποφάσει, λένε έχουμε ένα στόχο του 20%, 25-30% προ την Κομισιόν και του λένε κοιτάξτε να δείτε πόσο επιτυγχάνουμε αυτό το στόχο. Αναπόφευκτα, καταλήγουμε σε μια διαδικασία όπου η Επιτροπή θα δείξει κάποια γενοδορία προς τον εαυτό της ε, όσον αφορά τον υπολογισμό των δαπανών. Ένα νέο βελτιωμένο σύστημα θα χρειαστεί μια πιο αυστηρή προσέγγιση όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων, το μηχανισμό παρακολούθησης και τις πολιτικές αποφάσεις ε, όσον αφορά τους κλιματικούς στόχους ούτω ώστε να αντιμετωπιστεί το επίγον κλιματικό ζήτημα. Για τα μέλη που είπαν ότι οι δαπάνε για το κλίμα ενδεχομένω να μην έχουν τόσο μεγάλη προτεραιότητα λόγω τη κρίση του COVID, εγώ δεν θα συμφωνούσα απόλυτα. Κατά μία έννοια, δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες ε, που μας προσφέρονται για να διασφαλίσουμε καλύτερες δαπάνες ε, και ε, καλύτερες, ε, πιο πράσινες δαπάνες και μια πιο πράσινη οικονομία. Κοίταω τώρα τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Η κυρία Λαπόρτ νομίζω ειδικότερα ρώτησε τι γίνεται με τις διαφορές όσον αφορά την προσέγγιση του ΩΣΑ για την ε, για το fracking. Η προσέγγιση της ε, Κομισιόν ουσιαστικά είναι ε, μια προσέγγιση που συνάδει με το μηχανισμό που έχουμε προτείνει. Εστιάζεται στη συμβολή του προγράμματος για την επίτευξη των κλιματικών στόχων. Αντί λοιπόν να κοιτούν το σκοπό, κοιτάνε να δουν ε, αν οι δαπάνες έχουν αποτέλεσμα. και να μην είμαστε υπερβολικά γενναιόδοροι για κάποια από τα προγράμματα δαπανών. Ένα μέλος του ECR ρώτησε κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος λόγω της ε, εστιασμού στις κλιματικές δαπάνες το να στερήσουμε κάποια κρατημέλη από τις δυνατότητες ανάπτυξης. Είναι πολιτικό θεωρώ το ζήτημα, δεν θέλω να εμπλακώ σε τέτοια συζήτηση, εκτός το ότι να πω ότι η εστίαση στο κλίμα σε πολλές περιπτώσεις βοηθά την πιο αποτελεσματική ανάπτυξη των ε, κοινωνιών. Ο κύριος Κόκαλης ε, είπε ότι ήταν ανεπαρκές σε μεγάλο βαθμό το σύστημα της Κομισιόν. Είπε ότι είναι πολύ ε, θαραλέες οι λέξεις που χρησιμοποιούμε στην έκθεση. Φοβάμαι πάντα όταν με κατηγορούν ότι είμαι θαραλέος. Αλλά αυτό που θα έλεγα να πω είναι ότι πρέπει να προσέξουμε το πολιτικό βάρος που έχει ε, η παρακολούθηση του κλίματος αυτή τη στιγμή. Ε, καθώς το κλίμα αποτελεί όλο και πιο σημαντικό πολιτικό ζήτημα και η πολιτική κρίση γίνεται όλο και χειρότερη, ε, ο μηχανισμός που χρησιμοποιούμε για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσης γίνεται όλο και πιο σημαντική και εξού και η αυστηρότητα και η ακρίβεια αυτών των μηχανισμών γίνεται όλο και πιο σημαντική. Κύριε Λαρωτηρού, οι ερωτήσει σας αφορούσαν περισσότερο την Κομισιόν στράφηκε, ρώτησε εμένα κατά πόσο χρειάζεται ένα στιβαρό μηχανισμό σε τοπικό επίπεδο. Το υποστηρίζω. Πιστεύω ότι παίζει ζωτικό ρόλο να υπάρχει δράση σε τοπικό επίπεδο και οι σχετικοί φορείς να καταλαβαίνουν πώς ε, η δική του συμβολή ε, φέρνει ένα ευρύτερο παγκόσμιο αποτέλεσμα. Ο μηχανισμός παρακολούθησης ε, είναι υπερβολικά top-down και υπερβολικά γενικό και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να μεταφραστεί και στο τοπικό επίπεδο. Έχει δίκιο ο κ. Λορτουρού που εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι οι τοπικοί φορείς θα έχουν μια σαφή εικόνα του πώς συμβάλλουν και αυτοί τοπικά στην ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να μην μακρηγόρησα υπερβολικά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Νέσμπιτ, για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ κύριε Νέσμπιτ για τις απαντήσεις και ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές για τα σχόλιά τους. Ολοκληρώσαμε το σημείο 5 τη μέρης διάταξη για την εσωμάτωση τη διάσταση του κλίματο στον κοινοτικό προπολογισμό. Και περνάμε στι ψηφοφορίε, Πριν τι ψηφοφορίε όμω θα μα κάνουν μια ενημέρωση οι συγγητέ. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τι συγγητρίε. Ε, καταρχήν ε, για το τμήμα Μεταφορές 2020, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κυρία Χολμάιρ είναι η συγγετρία, είναι συνδεδεμένη η παρούσα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Also πρέπει να ρωτηθούμε Μόνικα. Κυρία Χολμάιερ, ε, καταρχήν είστε έτοιμοι να μας μιλήσετε, είσαι μένα τουλάχιστον. Α, φαντάζομαι πως είστε. Μόνικα, άναψε και την κάμερά σου. Γιατί αλλιώς μόνο γερμανικά θα σε ακούσουμε. Δεν έχει, προβλέπεται μετάφραση αν δεν υπάρχει και εικόνα. Μόνικα. Μόνικα. Hello. Can you hear me? Yes, I can hear you. you... Μ' ακούτε τώρα? Σας ακούμε. Δυστυχώς χωρίς εικόνα, κυρία Χολμάιερ, δεν μπορούμε να τη μεταφράσουμε. Translations, Monica. see everybody and hope that I see you soon in Brussels uh, um, again. Uh, Ελπίζω να τα ξαναπούμε και να τα αμώσουμε σύντομα στις Βρυξέλλες. Έχω ένα θέμα μόνο, πολύ σύντομο και σαφές. Πρόκειται για την μεταφορά DEC 15 του 2020 αφορά την ε, κινητοποίηση του αποθεματικού έκτακτης βοήθειας για να ανταποκριθούμε στη παροχή άμεσης, αποτελεσματικής και βάσει αναγκών ε, ανθρωπιστικής και πιστιστικής βοήθειας μετά από κάποια περιστατικά που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν όταν θεσπίσαμε τον προϋπολογισμό. Ε, συγκεκριμένα ε, αναφερόμαστε εδώ στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Λίβανο μετά τις καταστροφικές εκρήξεις στο λιμάνι της Βηρητού στις 4 Αυγούστου 2020. Ε, είχαμε 200 νεκρούς, πάνω από 6.000 τραυματίες και 600.000 ε, άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Έχασαν τις αιστείες τους, έχασαν τις επιχειρήσεις τους. Γι' αυτό και προτείνουμε ε, μεταφορά 30 εκατομμυρίων ε, σε πιστώσεις ε, πληρωμών και ενάλυψη υποχρεώσεων προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε κάποιες υγειονομικές παρεμβάσεις εκτάκτου ανάγκης, στέγαση, ίδρευση, αποχέτευση, πιστιστική βοήθεια, προστασία και παιδεία. Νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε την έγκρισή μας για αυτή τη μεταφορά. Μάλιστα. Και για το σημείο 6 μεταφορές 2020 για τα λοιπά τμήματα. Κυρία κυρία Γουαρδιασάβαλ Ρουμπιάλ είναι η εισηγητρία. Όπως είπατε έχουμε τέσσερα αιτήματα για μεταφορές. Η πρώτη προέρχεται από την Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή, αφορά περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Ε, η μεταφορά αυτή στόχο έχει να καλύψει τις ανάγκες επενδύσεων σε κτίρια και τεχνολογίες πληροφορίας όπως είπα, αφορά δημοσιονομικές γραμμές που κατά παράδοση ήταν υποχρηματοδοτούμενες από προηγούμενους προϋπολογισμούς και δοθεί σε ευκαιρίες ε, και μια και υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια σε άλλε δημοσιονομικέ γραμμέ, προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες προτείνοντα τη συγκεκριμένη μεταφορά. Και μάλιστα είναι σχετικά μικρή η δαπάνη λόγω και του κορονοϊού, της κρίσης, της πανδημίας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λοιπόν αυτοί τα 3 εκατομμύρια για να χρηματοδοτηθούν κτίρια και πληροφορική. Δεύτερη μεταφορά επίσης αφορά την Κοινωνική και Οικονομική Επιτροπή. Εδώ μιλούμε για 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Στόχος ε, της μεταφοράς είναι να υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα κονδύλια στον προϋπολογισμό για να γίνει μια προκαταβολή πληρωμών μισθωμάτων για του χρόνου και έτσι και στις επόμενες χρονιές ε, να υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο για χρηματοδότηση άλλων δαπανών και τα 5,5-7 εκατομμύρια θα προέρθουν από αντίστοιχες γραμμές ε, που χρησιμοποίησαμε και στην προηγουμένη μεταφορά που είχαν ε, υποεκτέλεση. Επίσης έχουμε 850.000 μεταφορά 5 του ελεκτικού συνεδρίου για να αυξηθεί μια δημοσιονομική γραμμή προκειμένου να βελτιωθεί η υποδομή για την αποθήκευση δεδομένων και θα προέλθει από τις αμοιβέ και ε, ημερήσεις αποζημιώσεις και η υπαριθμόν 6 μεταφορά του ελεκτικού συνεδρίου είναι 179.000 για την αγορά αδειών και χρηματοδοτικών χρηματοοικονομικών βάσεων δεδομένων και πρόσβαση σε κάποια online media. Ε, θα προέλθουν ε, από γραμμές για τις δημοσιεύσεις, την εκτύπωση δημοσιεύσεων μια και τώρα οι περισσότερες δημοσιεύσεις γίνονται επιγραμμικά και γι' αυτό έχουμε υποαπορρόφηση της συγκεκριμένης δημοσιονομικής γραμμής και υπάρχει διαθέσιμο κονδύλιο για μεταφορά. Αυτά νομίζω ότι έχετε λάβει όλες σχετικές πληροφορίες. Εγώ είμαι υπέρ ε, και των τεσσάρων μεταφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Από τους κοιόδους συζητητές, θέλει κάποιος το λόγο μήπως. Όχι από ό,τι βλέπω. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση αυτή. Όσον αφορά την ψηφοφορία αυτή αυτή, πρέπει να ελέγξουμε πρώτα απ' όλα την απαρτία. 11 ευρωβουλευτές. Για να ελέγξουμε λοιπόν. Ε, Παρακαλώ, αν ε, βρίσκεστε εξ αποστάσεως, πατήστε το κουμπί με το οποίο ζητάτε να παρέμβετε. Raise your hand. Και τους υπόλοιπους τους μετράμε εδώ στην αίθουσα. Ένας ακόμα. Έναν χρειαζόμαστε ακόμα. Α, είναι εδώ. Ναι, ωραία. Εντάξει, έχουμε απαρτία λοιπόν. Συνεπώς, ε, ζητώ Πρώτα απαρτία, επαληθεύτηκε. Τώρα, κατά τα άλλα, θα ψηφίσουμε τις τροπολογίες που έχουν υποβληθεί στην έκθεση όσον αφορά το σύστημα ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρεις γνωμοδοτήσεις. Πρόκειται για τα προγράμματα Health for You, React EU και την πολιτική προστασία. Οπότε η ψηφοφορία ξεκινάει τώρα μέχρι τις 16.45. Και έτσι εδώ ολοκληρώνεται η συνεδρίασή μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 1.45, 13 και 45, όπως ξεκινήσαμε και σήμερα δηλαδή. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας απόγευμα. this with me or do you want to take it with you? I'll take it with me because you have already a lot to...